Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε πολύ σημαντική μέρη σε διάταξη σήμερα και ήδη έχουμε δεκάλεπτη καθυστέρηση. Γι' αυτό μην χάνουμε άλλο χρόνο να ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε με το σχέδιο. Έχετε καμία αίσθηση, ο κύριος Βανίστερα. Όχι ακριβώς αίσθηση. Άρα είναι περίεργο ότι θα έρθει μετά την ψηφοφορία ο Επίτροπος. Ο κύριος Κατάινεν. Ναι, το δέχομαι. Τον είχαμε προσκαλέσει από το Φεβρουάριο, αλλά κολλιόταν τότε. Γι' αυτό και θα έρθει σήμερα τελικά. Δυστυχώς ε, θα έχει προηγηθεί η ψηφοφορία της ανταλλαγής απόψεων ε, με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με πάση περιπτώσει θα είναι χρήσιμη και ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων, παρόλο που γίνεται λίγο κατόπιν ε, εορτής, κατόπιν ψηφοφορίας. Άλλες παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη υπάρχουν, όχι, οπότε την εγκρίνουμε. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών. Τη συνεδρίαση της 26 Φεβρουαρίου. Το έχετε λάβει, οπότε Έχετε μέχρι το τέλος της συνεδρίας χρόνο να υποβάλλετε παρατηρήσεις, αλλιώς θα θεωρηθούν ε, εγκεκριμένα. Συμφωνείτε, πολύ ωραία. Σημείο 3, ανακοινώσεις της Προέδρου. Τρεις ανακοινώσεις μόνο έχω. Οι δύο είναι τεχνικής φύσεως και η τρίτη ενημερωτικής. Ανακοίνωση πρώτη Μην ξεχνάτε ότι στις 10 θα αρχίσει η ψηφοφορία. Φροντίστε να, να έχετε μαζί σας την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας, γιατί μερικές ψηφοφορίες θα γίνουν ηλεκτρονικά. Οπότε μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Ανακοίνωση δεύτερη. οι συνεδριές της Επιτροπής μας ε, στις 5 το απόγευμα. Δυστυχώς, φέτος, έχουμε πολλές ε, απογευματινές συνεδριάσεις ημέρα Πέμπτη. Και για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, όταν πρότεινα το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για όλο το χρόνο, περίμενα αντιδράσεις από εσά. Αλλά ούτε μία αντίδραση. Δεν άκουσα. Γι' αυτό και παγιώθηκε η πέμπτη το απόγευμα. Δεν έχουμε μόνο αυτή τη σημερινή, έχουμε άλλες τρεις απογευματινές της πέμπτης. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι συνεδριάσει της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις πέμπτες το απόγευμα γιατί πρέπει να διεκπαιρεώσουμε τις εργασίες μας και δεν προλαβαίνουμε μόνο με ένα πρωινό. Οπότε φροντίστε να ρυθμίσετε τα ταξιδιωτικά σας λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμά μας. Πάντως θα προσπαθήσω τουλάχιστον η κατανομή των σημείων στην ημερήσια διάταξη να γίνεται με δίκαιο τρόπο <coughs> ώστε όλες οι ομάδες να έχουν εξαίσθηση στις 5 το απόγευμα, γιατί ξέρω ότι τα απογεύματα είναι τα πιο δύσκολα. Το επιχειρήσαμε ήδη μία φορά, ε, να αλλάξουμε τελευταία στιγμή την ημερήσια διάταξη, δεν τα πολύ καταφέραμε, αλλά θα προσπαθήσω να φροντίσω μια, για μια δίκαιη κατανομή των θεμάτων ε, για την πέμπτη το απόγευμα, ώστε όλες οι ομάδες να έχουν εξαίσθηση και το πρωί και το απόγευμα. του χρόνου η Γραμματεία θα πιέσει ε, τις κεντρικές υπηρεσίες για μια καλύτερη κατανομή των ε, ημερών συνεδριάσεών μας. Γιατί πολλές άλλες επιτροπές δεν έχουν ε, πέμπτη απόγευμα συνεδρίες. Η κυρία Κρέλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ε, νόμιζα ότι είχε αλλάξει αυτό εκ των Δεν είχα προσέξει ότι υπήρχε τόσο συχνά συνεδρίαση το, την Πέμπτη το απόγευμα. Την άλλη φορά που θα το προσέξετε να μας το πείτε για να διαμαρτυρηθούμε γιατί προφανώς οι εργασίες στο Κοινοβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες είναι πολύ σημαντικές αλλά και στις ε, εκλογικές μας περιφέρειες είναι πάρα πολύ σημαντική η εργασία και έχουμε έτσι και αλλιώς μόνο την Παρασκευή και το Σάββατο και οι πιο πολλοί δεν μπορούν καν να φύγουν μετά τις 7 το απόγευμα την Πέμπτη. Ίσως μέσα στο Βέλγιο. Ίσως άντε και ο Λάμπερτ να μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Άντε και στην ε, Γαλλία. Αλλά όταν είναι κανείς από Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία δεν μπορεί να φύγει πιο αργά. Γι' αυτό λοιπόν δεν ε, είναι δυνατόν γίνεται και με τους αναπληρωματικούς που αναπληρώνουν τα, τα μέλη που λείπουν. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να το αποφύγουμε αυτό σε μια συζήτηση, σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία. Θα πρέπει να είναι δυνατό να οργανώνει, ε, να η κάθε ομάδα προκειμένου να υπάρχει ένας τουλάχιστον ομιλητή. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τα σχόλιά σας. Έχουμε και εμπειρία από την προηγούμενη συνάντηση άλλωστε η κατάσταση αυτή με τις ε, απογευματινές συνεδριάσεις της Πέμπτες ίσως να μας οθήσει με καλό τρόπο να είμαστε και πιο ευέλικτοι για να αποδεχόμαστε τα άτομα που αντικαθιστούν κάποιους συναδέλφους τους. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα αυτό. Το καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω. Να φύγει κανείς για να πετάξει για Βουλγαρία από εδώ. Άρα αναγκαστικά χάνω όλη την Παρασκευή γιατί πρέπει να πάρω μια πτήση Παρασκευή πρωί. Αλλά έτσι έχει η κατάσταση με τις συνεδριάσεις μας. Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση, να οργανώσουμε λίγο την ατζέντα μας και το χρόνο εργασίας μας και αναλόγως και τις πτήσεις μας. Να προσπαθούμε να βρούμε άτομα να μας αντικαθιστούν σε κάποιες συνεδριάσεις και να διαβεβαιώσουμε ότι, να εξασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας εδώ στην Επιτροπή. Θα κάνουμε κάτι καλύτερα για τον χρόνο, ελπίζουμε. Τρίτη ανακοίνωση τώρα από την Πρόεδρο. Σας ενημερώνω ότι την προηγούμενη εβδομάδα προείδρευσα μια αντιπροσωπεία ε, της Επιτροπής Ρέτζης στις 100 ε, χώρες. Η πρώτη αντιπροσωπεία, η πρώτη μάλλον αποστολή και αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Τα άλλα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν η κυρία Γκουεφρίδα, κύριε Μαζέ, Νοβάκοφ, η κυρία Ντροτρίκες και η κυρία Σπυράκη. Ο κύριος Πανίστελ Ροή μας συνόδευσε. Να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την υποστήριξή του και την υποστήριξη του γραφείου του στο πρόγραμμά μας και στις επισκέψεις μας. Μείναμε εντυπωσιασμένοι από τις συνεδριάσεις στις κάτω χώρες. Ήταν πολύ θερμή υποδοχή και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και επικοδομητικές οι συνεδρίσεις μας. Είμαι βέβαιη ότι αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς η περιφερειακή πολιτική και ο αντίκτυπος του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιφέρει ανάπτυξη για θέσεις απασχόλησης και πρόοδο, εξελίξεις ε, για την τοπική οικονομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αποστολής μας ήταν να συμμετάσχουμε σε μια εξαιρετικά καλή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, των τοπικών περιφερειακών αρχών, των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών επιστημονικών ιδρυμάτων. Όλα αυτά εγγυώνται μια καλή εξέλιξη σε οποιοδήποτε έργο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κύριε Φανίστολ Ροή. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή. Θα ευχαριστήσουμε και επίσημα όλους αυτούς που μας υποδέχτηκαν, επιχειρήσεις, οργανώσεις, ευρήματα. Με μεγάλη επιτυχία λοιπόν στέφτηκε αυτή η πρώτη αποστολή. Θα συζητήσουμε και στις επόμενες αποστολές για την φετινή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων και την πολιτική συνοχή και αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ευρώπη 2020. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Ρούα. Είναι εδώ. Έχουμε και σκιώδεις εισηγητέ, εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί μα. Είναι τον κύριο Μαρσέλ Χάρκ και την κυρία Αλβάν Τίμπλα από τη Γενική Γραμματεία και τον κύριο Τζον Βόλς από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Όντω έτσι, στέκει αυτό, μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Ρούα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια διπλή μου ιδιότητα για 24 χρόνια ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μιας πόλης της Πρωτοβουλής και τελευταία δύο χρόνια πρόεδρος της ε, Ένωσης ε, Πρωτογαλλικών Δήμων. Γι' αυτό αισθάνομαι τεράστια ευθύνη ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της Επιτροπής και της έκθεσης που έχω αναλάβει. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Έχουμε τώρα μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων της έκθεσής μου, που είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Θέλω να ακούσω τα δικά σας σχόλια και να σας διαβεβαιώσω για την προθυμία μου ε, να εμβαθύνουμε τις επόμενες εβδομάδες τη συζήτηση, να έχουμε πολλές συνομιλίες, είτε διμερείς, είτε άτυπες, είτε επίσημες. Στόχος μου είναι να συντάξω μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για την πολιτική συνοχής ε, εν ώψη της μεταρρύθμισης ε, της ε, πολιτικής Ευρώπη 2020. Θέλω να είναι δυναμική έκθεση, περιεκτική και να συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γίνει δικαιότερη και ισχυρότερη αυτή. Θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται η έκθεση. Όπως θα γνωρίζετε, και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχουν δημοσιεύσει τις ιστοσελίδες του σχετικά έγγραφα για τη διαδικασία της ενδιάμεσα αναθεώρησης ε, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μάλιστα για το πρώτο εξάμεινο του 2015 είχε αναγγελθεί η υποβολή αυτής της ε, ενδιάμεσης αναθεώρησης. Και, και η ΟΚΕ και η Επιτροπή Περιφερειών ε, έχουν συντάξει γενικά τους έγγραφα και υπάρχει και μια μελέτη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ε, που εξετάζεται αυτή τη στιγμή με τους εταίρους. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5 Μαρτίου του προηγούμενου έτους ε, εγγενίασε δημόσιες διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αυτή αναθεώρηση και μάλιστα αυτό το μήνα είχαμε και τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. Στην ανακοίνωση του Μαρτίου, του προηγούμενου Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι η πρότασή τη για την ενδιάμεση αναθεώρηση θα υποβληθεί στα τέλη του έτου με βάση το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015. Ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Καϊτάνα, ε, είπε το Φεβρουάριο ότι δεν έγινε υποβολή αυτό το εξάμεινο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την ανάλυση της κατάστασης αλλά και για την ικανοποίηση άλλων προτεραιοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι το γενικότερο πλαίσιο και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή θα εξετάσουμε αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για την πολιτική συνοχή στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Εγώ θα σας εξέσω εδώ πέντε βασικές ιδέες για την έναρξη της συζήτηση και περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις, σκέψεις, προτάσεις και ιδέες. Θεωρώ καταρχήν ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε τον κεντρικό και ζωτικό ρόλο της πολιτικής συνοχής για την έμπρακτη εφαρμογή των μέτρων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεύτερη ιδέα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ταμείο δηλαδή και τα ταμεία του σχεδίου Juncker, θα πρέπει να συμπληρώνουν την πολιτική σχέση και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία τα υπάρχοντα. Τρίτη ιδέα. Η στρατηγική 2020, Ευρώπη 2020, θα πρέπει να στηρίζεται σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με βάση την αρχή της εταιρικότητας, της εταιρικής σχέσης. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε μια μεικτή προσέγγιση και από τη βάση προς την κορυφή και τα ναπαλιν Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που ήδη εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Για να ελαχιστοποιήσουμε τη, τον κίνδυνο υπερφόρτωση διοικητική των διαφόρων ε, επιπέδων τη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα των χαμηλών επιπέδων, θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να προωθήσουμε τη διοικητική απλοποίηση, αλλά να δώσουμε έμφαση στο θε, στη θεματική ενότητα 11, δηλαδή την ενίσχυση των διοικητικών ικανότητων. Τέταρτον, ανάγκη εδαφικής ε, προσέγγισης για την Ευρώπη 2020 να έχουμε μέτρα και στόχους ε, που θα προσαρμόζονται στις διατερότητες κάθε περιφέρειας, δηλαδή ειδικού ε, και εξατομικευμένους στόχους για κάθε περιφέρεια. Και είμαστε ε, βέβαια υπέρ της ευελιξίας ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των στόχων, για παράδειγμα μέσω αναλύσεων και ποσοτικών αξιολογήσεων. Είναι προφανές ότι οι διάφορες περιφέρειες έχουν διαφορετικά βιώματα, διαφορετική πραγματικότητα και ιδιαιτερότητες το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, σίγουρα θα αυξήσουν την αίσθηση της ιδιοκτησίας της στρατηγική του Ευρώπης 2020. Δηλαδή, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα κάνουν κτήμα τους στους στόχους αυτής της αρχής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα συμβάλλουν έτσι και οι τοπικές αρχές πολύ καλύτερα. να θεωρήσουν κτήμα τους αυτή την ε, στρατηγική στην υλοποίηση των στόχων τη Δεδομένων ε, των χρονικών περιορισμών και των καθυστερήσεων που έγιναν στην περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, θεωρώ ότι η συζήτηση για τα μελλοντικά διαρθρωτικά ταμεία και τη μελλοντική μακροπρόθεσμη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για το επομενο πολιτε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ε, η αναθεώρηση της ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να γίνει με σταδιακό τρόπο και περιεκτικό για να αποφευθούν τα λάθη του παρελθόντος και να εφαρμοστούν και εμπράκτως οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι από το 2019 θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε θα ασχοληθούν όχι μόνο με την αξιολόγηση της υφιστάμενης στρατηγικής Ευρώπη 2020, αλλά θα έχουν την ευθύνη να χαράξουν και μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να θεσπίσουν και ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με βάση το, το νομοθετικό πλαίσιο. Να σας υπενθυμίσω και το χρονοδιάγραμμα της έκθεσής μου. Στις 17 Ιουνίου θα έχουμε τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και την εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Τον Ιούλιο ε, θα λήξει προθεσμία για τις τροπολογίες και τις 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω την ε, ανυπομονησία μου και την προθυμία μου να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ, Λεπρόεδρο, για το δώσουμε το λόγο στους και ηγητές. Η κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ και για την ε, δυνατότητα που μας δίνετε σε μια πρώτη που μας δώσατε μάλλον σε μια πρώτη συνάντηση των σκιωδών να κάνουμε μια σχετική συζήτηση. Κάτι ερωτήσει <coughs> έχω να κάνω. Είναι εξαιρετική η έκθεση και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα σημεία τα οποία ανέφερε και ο εισήγητής. Υποστηρίζω ξεκάθαρα το γεγονός ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τους στόχους για το 2020 με την πολιτική συνοχή, γιατί η πολιτική συνοχή είναι το κατεξοχήν εργαλείο για την εφαρμογή της στρατηγική αυτής. Και αν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες θέλουν να πετύχουν τους στόχους αυτούς, θα πρέπει να εργαστούν προφανώς και με την πολιτική συνοχή. Αυτή είναι η λογική. Υποστηρίζω επίσης ε, τα σημεία τα οποία ανέφερε ο εισηγητής για τις εταιρικές σχέσεις και τη σχετική στρατηγική. Θέλουμε μια αρχή εταιρικής σχέσης καλύτερα διατυπωμένη. Το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ και ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι οργανωμένα στις περιφερειές όπως αρχικά σκοπεύαμε. Και εκ των υστέρων προφανώς δεν θα έχει μεγάλο νόημα να διακόψουμε τη διαδικασία και να αλλάξουμε την αρχή εταιρική σχέση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να το αποδεχτούμε έτσι απλά και ότι η μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει ανάλογα να προωθηθεί. Θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό στην επόμενη περίοδο. Το θέμα των περιφερειακών στόχων, σημαντικό σε κάθε περίπτωση, αλλά να παρακαλέσω τον εισήγητη να βρει μια σωστή διατύπωση στην έκθεσή του, γιατί θα πρέπει να προσέξουμε στους ευρωπαϊκούς στόχους, στους εθνικούς στόχους, στους ε, περιφερειακούς στόχους που θα πρέπει να ελεγχθούν και έτσι θα προκληθεί γραφειοκρατικό άχθος, το οποίο δεν επιθυμούμε. Εμεί είμαστε υπέρ της μείωσης του γραφειοκρατικού κόστους και άχθους. Άρα η προσθήκη ενός επιπρόσθετου επίπεδου στόχων θα μπορούσε, θα μπορούσε λέω, να οδηγήσει σε επιτείνωση της κατάστασης για τις ε, περιφέρειες και τους ε, δήμους. Σίγουρα δεν ε, θέλει να πετύχει αυτό ο εισηγητής. Χαίρομαι που ανέφερε το σχέδιο σε ο εισηγητής και την προετοιμασία της επόμενης περίοδου. Δύο φράσεις να πω όμως, δύο προτάσεις επιτρέψτε μου. Στην τελευταία θητεία, στο 2010, ξεκινήσαμε να συζητάμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική συνοχή για την ψήφιση του κανονισμού που τελικά ψηφίστηκε το 2014, το Δεκέμβριο, το 2013. Δεκέμβριο 2013, διαφωνεί η ομιλήτρια, για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Δεν τα καταφέραμε. Γιατί αυτόν τον κανονισμό τελικά αναγκαστήκαμε να τον ε, διαπραγματευτούμε σε πάνω από 100 τριμερείς ε, διαλόγους. Θα ήταν καλύτερο να υπήρχε μεγαλύτερη και πιο αποδοτική συνεργασία με το Συμβούλιο ή μάλλον το Συμβούλιο να συνεργαστεί καλύτερα μαζί μας γιατί εμείς τελικά πατήσαμε το φρένο. δεν υπήρχε μεγάλη ευελιξία, αλλά αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και το ξέρω αυτό, που μπορούμε να το πετύχουμε από, το, από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Μπορούμε ήδη να ζητήσουμε μια συζήτηση για, την, για τον καθορισμό κάποιων δικτών που το είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά. Αν αυτό μπορούμε να το οργανώσουμε τώρα και να το συμφωνήσουμε, έχουμε ένα μεγάλο χρονικό περιθώριο το οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για άλλους σκοπούς. Και θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε τι δείκτες χρειαζόμαστε για την επόμενη πολιτική συνοχή προκειμένου να είναι και μετά το 2020 αποτελεσματική πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κρέλη. Η πρόεδρος δίνει το λόγο στην κυρία Τόμασιτς. Αλλά απουσιάζει. Φαν Μίλτενμπουργκ. Σκιώδης ηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή, όπως υπόθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020. Καθοριστικό, λοιπόν, εργαλείο. Και για την ε, Ένωση Καινοτομία, εμβληματική πρωτοβουλία για την ε, Ευρώπη του 2020, όπου η πολιτική συνοχή μπορεί να συμβάλλει προκειμένου να υπάρξει βελτιστοποίηση κοιτώντα τον αντίκτυπο, μάλλον τα αποτελέσματα της, της διαβούλευσης, της δημόσιας διαβούλευσης που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη 2020, διαπιστώνουμε ότι το 2013 είμαστε στο 2% περίπου σε ό,τι αφορά το μερίδιο του ΑΕΠ για τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να είμαστε γύρω στο 3% σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη που μπορούν θεωρούμε να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης άρα. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, τα κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο κυρίως μπορούν να προοριστούν και να δαπανηθούν στην ε, ατζέντα για το ανθρώπινο δυναμικό. Ένα άλλο σημείο. Πώς θα ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς θα ενισχύσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλα αυτά τα ζητήματα μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020. Θεωρώ ότι είμαστε σε σωστό δρόμο με τα πλαίσια τα οποία έχουμε δημιουργήσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα άλλα θεσμικά όργανα στην πολιτική συνοχή, αλλά ξέρουμε ότι τώρα σιγά σιγά θα πρέπει να εγκρίνονται σιγά σιγά αυτά τα προγράμματα. Τώρα λοιπόν έχουμε περάσει στην φάση της εφαρμογής, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε τα κονδύλια τα οποία δαπανούνται από την πολιτική συνοχή να έχουν αποτέλεσμα και αντίκτυπο για να πετύχουμε την ε, στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Ε, θα περιγραφώ λοιπόν σε αυτά και ελπίζω να τα λάβει υπόψη αυτά ο εισηγητή. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, πρόεδρο. Ο επόμενο πιο εισηγητή είναι ο Δημήτρης Παπαδημούλη. Αλλά δεν είναι εδώ. Uh, You don't want. Okay. Okay. Α, δεν θέλετε να μιλήσετε εσείς. Καλά. Mr. Rope, will you take the floor? Κύριε Ρόπε, θέλετε το λόγο. Ορίστε. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή Λυκής Ροπέ. Εγώ έχω προεδρεύσει ενός φορέα δημάρχων στην ε, Λιθουανία και έχω κάποια ιδέα για το πώς λειτουργεί η πολιτική συνοχή στα κράτη-μέλη. Θα συμμετάσχω σε όλες τις ε, συναντήσεις που θα γίνουν με τους κοιόδης ηγητές και Νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη που τα πράγματα είναι καλύτερα και που είναι λιγότερο καλά. Χθες συζητήσαμε για τα προβλήματα στις μεταφορές στην Ευρώπη και είπαμε ε, τι γίνεται με την ελάχιστη αμοιβή, τον ελάχιστο μισθό στην Γερμανία και είδαμε πόσα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάποια κρατημέλη. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε ε, αυτές οι διαφορές ε, κάπως να γεφυρωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω θα πρέπει το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων να λειτουργεί αποκεντρωμένα και έτσι να βοηθήσει στο να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε μια πραγματική συνοχή. Λέει ο εισηγητής μεταξύ άλλων ότι έχουμε διακυβέρνηση πολυεπίπεδη και αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται φυσικό το τρόπο. Έχουμε εμπειρία σε αυτό το τομέα γιατί η Λιθουανία επειδή είναι μικρή χώρα θεωρείται περιφέρεια, μία περιφέρεια και επομένως είχαμε ηγετικό ρόλο ας πούμε στην αντιμετώπιση της περιφερειακής πολιτικής άρα θα πρέπει όλα τα κρατημέλη να εφαρμόσουν μια περιφερειακή πολιτικης αρα θα πρεπει ολα τα κατημέλη να εφαρμοσουν μια περιφερειακη πολιτικη και να μην μείνουμε στα λόγια να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο κάποια στιγμή να εφαρμοστεί, οπότε θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη και οι φορείς οι περιφερειακοί. Να συνοηθούμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει επομένως δήμοι και κοινότητες να εμπλακούν περισσότερο, να έχουν περισσότερα δικαιώματα και αρμοδιότητες και έτσι θα βγουν όλοι κερδισμένοι. Γιατί οι δήμοι και κοινότητες ενδιαφέρονται για τις επενδύσεις που θα βελτιώσουν την ε, περιοχή τους. Και τα πολιτικά κόμματα όλα θα ενδιαφερθούν και όλοι θα βοηθήσουν να ελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Επομένως θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη μιας περιοχής. Επομένως, ε, οι, οι τοπικές αρχές πρόκειται να ασχοληθούν μετά του τόπου τους, δεν χρειάζεται να αναμειχθεί ε, η κεντρική εξουσία, ε, δεν χρειάζονται φορολογίες και τέτοιου ισοδύναμα μέτρα. Στη Λιθουανία 11% των πόρων πήγαν στην περιφερειακή πολιτική. Οι υπόλοιποι όλοι πόροι έμειναν στο κέντρο, στην κεντρική εξουσία. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, κατά τη γνώμη μου. Τουλάχιστον το μισό αυτών των πόρων θα πρέπει να κατευθυνθούν προς δήμους και κοινότητες και εκείνοι να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Στην αρχή κάθε περίοδου προγραμματισμού βλέπουμε νέους κανόνες. Οι δε τοπικές αρχές χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους και ε, τρέχουν ούτως υπήν τα, το 70% των projects και σχεδίων. Πρόεδρος και τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να, να μιλήσουν έχουν μέρο στην συζήτηση. Έχει δει κάποιο το λόγο. Ο κ. Φανή Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μια βάση κίνηση για αυτή τη συζήτηση και έχω να παρατηρήσω τα εξή. Τώρα προσέρχεται μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα έκανε την αξιολόγηση για το 2016. Και λέμε ότι τώρα με αυτή την πρωτοβουλία μπορούμε να στιάσουμε την προσοχή μας στον ορίζοντα του 2020 και όλοι λέμε, όλοι εμπλεκόμενοι ότι καλά πάμε και είναι αυτό βασικό πιο πράσινο με μεφή τρόπο κλπ. Όμως τώρα θα πρέπει να δούμε τι μέσα πολιτικής έχουμε, τι μας προσφέρει ο κανονισμός και επί τη βάση αυτών αποδίδουμε τα πάμε καλύτερα από ό,τι στην προηγούμενη ε, περίοδο με τη στρατηγική της Λισαβόνας με τους παλαιότερους κανονισμούς. Τώρα έχουμε το 2020, έχουμε θεματική συγκέντρωση, νέους κανονισμούς. Να μην γίνει διασπάθηση των πόρων. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά χρήματα, οι ευρωπαϊκοί πόροι να πάνε στους συγκεκριμένους στόχους για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε εδώ κάποιους δείκτες που κυριαρχούν σε αυτό το σύστημα. Επομένως, θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο και να δούμε με τι σύστημα θα αποδώσουμε. Να μην τα κάνουμε τα πράγματα βουνό και δύσκολα. Μην τα κάνουμε γραφειοκρατικά. Ας ξεκινήσουμε από το ποιους στόχους θέλουμε εν ώψη του 2020 να πετύχουμε. Άρα ε, ας κάτσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να προετοιμαστούμε και στην Επιτροπή μας ε, ενημερωνόμαστε, συζητούμε, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε υπόψη ότι τα πράγματα μεταβάλλονται, μεταβάλλονται πάρα πολύ. Και μιλώ για ε, θέματα και εκτός περιοχής πολιτικής. Άρα θα πρέπει και στην Επιτροπή μας να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. και πάντοτε να έχουμε στο μυαλό πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Επομένως, περισσότερος χρόνος χρειάζεται. Συζητείτε το θέμα επίσης και στην Οικονομική Επιτροπή, σε όλο το Κοινοβούλιο θα, γίνει αυτή η ζήτηση του χρόνου. Έχουμε τώρα αυτή τη δική μας πρωτοβουλία και επομένως ας βρούμε τον χρόνο ούτω ώστε να προσαρμόσουμε κάποιες ε, ιδέες μας οι οποίες θα αξιοποιηθούν αργότερα. Mr. Van Nistelrooy, Madame Grazie, Presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μπρέσο. Έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα συζητήσουμε επί τη βάση του κειμένου που θα μας παρουσιάσει ο συνάδελφος. Θεωρώ ότι ως προπαρασκευή, ακριβώς όπως τονίστηκε, Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει πρόγραμμα και δράσεις για το, το Ευρώπη 2020, οπότε θα πρέπει να μας παρουσιάσει μια ανάλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κρίση. Γιατί το Ευρώπη 2020 ε, προέκυψε πριν την κρίση και έχουμε τώρα αυτή την κρίση που μας στείλει την Ευρώπη και οικονομική και κοινωνική και επομένως δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι εδώ πέρα πρόκειται για κάποιο είδου αναθεώρηση ρουτίνα. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Να κρατούμε και να αναλύσουμε το κατά πόσον οι στρατηγικές μας έχουν ή δεν έχουν την αναγκαία ευελιξία ούτω ώστε να προσαρμοστούν στην μεταβολή των πραγμάτων, στη μεταβολή της οικονομίας, του κόσμου, της κοινωνίας. Οπότε δεν γίνεται να μείνουν άκαμπτες οι στρατηγικές μας όσο και να συμφωνούμε γιατί θα, θα πρέπει να έχουν περισσότερη ε, ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής στην πραγματικότητα γιατί η Ευρώπη βασίζεται στον προγραμματισμό αλλά θα πρέπει οι λεπτομέρειες αυτού του προγραμματισμού να έχουν την ικανότητα προσαρμογής στην πραγματικότητα αλλιώς ο προγραμματισμός δεν θα αποδώσει. Όπως ξέρουμε ιστορικά να γίνεται. Και οι στόχοι θα μείνουν όνειρα σε εισαγωγικά. Άρα ευελιξία και προσωμή στην πραγματικότητα. Οπότε παρακαλώ τον συνάδελφο να απευθυνθεί στην Επιτροπή που για να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια όσον αφορά αυτού του είδους την διάρθρωση για τον προγραμματισμό των ε, βασικών στρατηγικών. Thank you. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Η κυρία Τόμασιτς. Καταρχήν σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήμουν σε τριμερή διάλογο στην Επιτροπή Αλίας. Αυτά από αγγλικής πλευράς, τώρα θα περάσω στα κρατικά. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 ξεκίνησε για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση πόρο ακόμη απέχουν από την υλοποίηση των στόχων τη στρατηγική. Εξαιτία τη μακροχρόνια οικονομική κρίση και τη μείωση των δημοσίων επενδύσεων, πολλέ περιφέρειε δεν μπόρεσαν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων τη Ευρώπη 2020. Και, ε, και 75% των ε, ε, των κατοίκων δεν μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτέ. Και μάλιστα η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ έπρεπε από τη στρατηγική, 2020 να τη χρησιμοποιήσουν ω γνώμονα τη δική του ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τι βέλτιστε πρακτικέ. Τα προγράμματα εθνική μεταρρύθμιση των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την υπερπίδηση των εμποδίων προκειμένου να έχουμε ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη δεν λαμβάνει υπόψη τις ε, τοπικές περιφερειακές ανισότητες και ιδιαιτερότητες ή τις, ε, τα τοπικά και περιφερειακά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. αναφέρεται η, η προσέγγιση ε, από την κορυφή προς τη βάση που περισσότερο χρησιμοποιήθηκε. Έμειναν πολλές αναξιοποιητές δυνατότητες. Ε, θα πρέπει να βελτιωθεί καλύτερη συνεργασία στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια συνδυασμένη προσέγγιση από την βάση προς την κορυφή και αντίστροφα και όχι μόνο από την κορυφή προς τη βάση. Με μια τέτοια διπλή προσέγγιση θα ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες και όχι μόνο η υλοποίηση των στόχων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια έτσι αναθεωρημένη στρατηγική θα συμβάλλει καλύτερα σε ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα καταστήσει πιο αποτελεσματικές και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ευχαριστώ. Before. ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επισέλθω... Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, κάποια γενικά σχόλια να κάνω. Και μια παρατηρήση που θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική όταν θα μιλήσουμε για το 2020. Η στρατηγική 2020 σημαίνει ότι δημιουργούμε μια ανάπτυξη και έτσι και θέσεις απασχόλησης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι περιφέρειες, ε, οι δήμοι να έχουν δυνατότητα να επενδύουν, να παίρνουν δηλαδή χρήματα στα χέρια τους και να πραγματοποιούν έργα να επενδύουν σε τέτοια ευφύη προγράμματα και έργα. Αυτό φυσικά με τα κριτήρια τα οποία έχουμε ορίσει στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, στο Six Pack, στο Two Pack. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνος που αναφέρω τα στοιχεία αυτά, ότι οι Δήμοι, τα κρατήδια, οι περιφέρειες έχουν τεράστιο πρόβλημα να επενδύουν σε έργα για το μέλλον. Θα πρέπει το πρότυπο, το οποίο είναι γνωστό και ως ΣΕΚ 2010, να φροντίσουμε να μην παρεμποδίζει τις επενδύσεις. Θα το συζητήσουμε αυτό λοιπόν στους κόλπους του Κοινοβουλίου. Δεν ε, είναι δική μου αυτή η παρατηρήση μόνο, γιατί αν μείνουν τα πράγματα Μα έχει αυτή η κατάσταση. Δεν θα μπορούν να υπάρχουν επενδύσει τόσο στο μέλλον. Γιατί είναι τεχνικά τα προβλήματα της απόσβεσης. Ακόμα και αν πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο στρέφεται στο μέλλον για ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να αποτυπωθεί κάπου γιατί αν δεν μπορούν τελικά να επενδύσουν τα κρατήδια, οι περιφέρειε, οι δήμοι, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο, η κυρία Μάλετσεβιτ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με του συναδέλφους ότι είναι πολύ δύσκολο ε, μεσούς της κρίσης να εξασφαλίσουμε μια δυναμική σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, αν δεν αλλάξουμε σημαντικά και το, την προσέγγιση μας και, το, και τη μεθοδολογία μας. Και είναι σημαντικό να δούμε τι συνέβη στην πολιτική συνοχής. Έχει αλλάξει η προοπτική που είχαμε το 2013 σε σχέση με τη νέα προοπτική που έχουμε και το 2014-2020. Και δεν άλλαξε μόνο η επενδυτική πολιτική, αλλά άλλαξε και η αναπτυξιακή μας πολιτική, προκειμένου να υλοποιήσουμε καλύτερα τους στόχους ε, της Ευρώπης 2020. Βέβαια, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και την όλη θετική και να αξιολογήσουμε το, τους στόχους της. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, και επίκαιρο να ασχοληθούμε με την αναθεώρηση αυτή τώρα, ώστε μέχρι το 2020 να έχουμε απτά και θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόλς είναι ο επόμενος ομιλητής. Here? Δεν είναι εδώ. Δεν θα είναι δεν θα μιλήσει ο κύριος Βούλς, είμαι από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, δηλώσεις αυτές. Πρόκειται για θέματα τα οποία τα εξετάζουμε για την ε, αναθεώρηση της ε, στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Όλα όσα ακούσαμε σήμερα σίγουρα θα επηρεάσουν και τις προπαρασκευαστικές μας εργασίες για την αναθεώρηση αυτή. Να πω δύο λόγια για τις πρόσφατες εξελίξεις για την ε, στρατηγική 2020 και το πώς συνδέεται με την πολιτική συνοχή. Το αναφέρατε σε διάφορες δηλώσεις και εσείς. Έχουμε προλιάνει το έδαφος, κάναμε μια διαβούλευση για να καταγράψουμε που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο για τους στόχους του 2020. Μετά ξεκινήσαμε τις δημόσιες ε, διαβουλεύσεις που αναφέρατε μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2014 και θα προχωρήσουμε σε δύο βήματα, σε δύο επίπεδα. Από 1η Μαρτίου 2015 θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης μαζί με μια ενημερωμένη έκθεση για το πώς έχει η κατάσταση για, την, στόχου τους στόχους της στρατηγικής αναχώρα. Λάβαμε πάνω από 700 απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση και το βασικό μήνυμα το οποίο τονίστηκε στις διάφορες δηλώσεις ήταν ότι γενικά η στρατηγική είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά τους στόχους για την επίτευξη θέσεων απασχόλησης, ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και ενδεχομένως να αντιμετωπίσει αύριο, ότι οι στόχοι για τις επικεφαλίδες είναι σωστοί και επιβεβαιώνουν και υποστηρίζουν οι μεν τους δε. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ανέκυψε ως αδυναμία της στρατηγικής από τις απαντήσεις, το αναφέρατε και εσείς, η ανάγκη να συμμετέχουν πιο πολύ διάφοροι φορείς, όχι μόνο οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στρατηγική. Να υπάρχει δηλαδή η ανάγκη να νιώθουν οι διάφοροι φορείς, οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς, ότι τους ανήκει, είναι δική τους αυτή η στρατηγική. Η δεύτερη φάση λοιπόν θα, θα θεωρήσει θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλη του 2015, οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει προτάσεις για την αναθεώρηση της στρατηγικής, γιατί στη δημοσίευση της ε, την 1η Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει ακόμα συμπερα... δεν έχει κάνει ακόμα συστάσεις. Πρόκειται ασφαλώς ε, για μια σημαντικότατη στρατηγική, ένα σημαντικότατο εργαλείο για την επιλέξη τη Στρατηγική του 2020 και οι τοπικές αρχές τη περιφερειακή αυτοδιοίκησης έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν σε ό,τι αφορά την επιτεύξη των προτεραιοτήτων για την Ευρώπη 2020. Αυτό που ανέκυψε ως αποτέλεσμα των αναλύσεων και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην αναθεώρηση είναι οι μεγαλύτερες αποκλήσεις, οι αυξανόμενες αποκλήσεις, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις εντός των διαφορετικών κρατών μελών. Μία κάποια αύξηση, λοιπόν, λόγω της κρίσης, των ε, περιφερειακών διαφορών στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών. Θα σταματήσω εδώ και ίσως θα ήθελα να πάρει ο συνάδελφος το λόγο για να συμπληρώσει τα όσα είπα. Η πρόεδρος. Κύριε Γουόλς, να σας δώσω το λόγο, αλλά να είστε πάρα πολύ σύντομος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω δύο λόγια για αυτά τα οποία παρουσίασε ο εισηγητής. Ναι, είναι πολύ αξιόλογη αυτή ως αφετηρία. Συμβάλλει αυτό στο έργο μας και νομίζω ότι πάρα πολλά από τα σημαντικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής έχουν προέλθει σαν ιδέες, σαν έμπνευση από τη στρατηγική 2020. Να σταθούμε σε δύο-τρία από αυτά τα σημαντικά σημεία. Εμείς μελετούμε το πώς αυτά τα καινούργια ενισχυμένα στοιχεία ε, έχουν ενταχθεί στην έκθεση και θα έχουμε κάποια έκθεση και εμείς ε, για την έκφραση των διαπραγματεύσεων. Και ε, από ό,τι άκουσα από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ότι είναι μια δοκιμή της της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης η πολιτική της συνοχής και με τον κώδικα διοντολογίας ενισχύθηκε και κινητοποιήσαμε τη συνδιαχείριση με τα κράτη-μέλη και του, τις τοπικές αρχές και άλλους εμπλεκομένους για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της ε, πολιτικής αυτής η οποία τώρα είναι πιο σωστά εστιασμένη και σε σχέση με την θεματική συγκέντρωση αλλά επίσης Έχουμε τώρα έναν πιο σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα σε σχέση με κράτη-μέλη και περιφέρειες, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιους ε, στόχους ε, καθορισμένους στα πλαίσια της διαδικασίας προγραμματισμού εν ώψη του 2020 και έχουμε αντιλήσει μαθήματα για το πώς θα γεφυρωθούν τα χάσματα και πώς ε, περιφέρειες και κράτη-μέλη ε, θα, θα, προσεγγίσουν την επίτευξη των στόχων. Εδώ βάλω μια τελεία και οπωσδήποτε θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας αλλά και το, βέβαια τον συντονιστή πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Ρούας, μήπως θέλετε το λόγο για τα τελικά σχόλια πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Λακωνικότατα κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέρφους ε, για τις παρατηρήσεις τους. Ε, τις ε, κατέγραψα, για παράδειγμα, απλούστευση και ελάφρυση του διοικητικού φόρτου. να δοθεί περισσότερη εξουσία στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εννοείται ότι οι τοπικοί φορείς με την Ευρώπη 2020 κάνουν πολύ περισσότερες επενδύσεις από ότι οι εθνικές αρχές. Είναι εκείνη η πραγματικότητα. Επίσης, ε, διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι οι προσανατολισμοί του προγραμματισμού θα πρέπει να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα. Και επίσης, τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για να τροφοδοτούν την οικονομία, αλλά και για να τη μετασχηματίζουν Ευχαριστώ λοιπόν ε, για την ευκαιρία της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Ε, πολύ επικοδομητική συζήτηση. Έχω καταγράψει τις παρατηρήσεις και ας μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, που δεν χαρακτηρίζεται όμως από σημαντικές ιδεολογικές διαφωνίες Γι' αυτό πιστεύω θα καταλήξουμε σε ένα κοινό παρανομαστή, σε κοινά σημεία που θα χαρακτηρίζουν την έκθεση. Ευχαριστώ. Μας αναφέρατε και το χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικές ανταλλαγές απόψεων, τη διορία ε, για τις τροπολογίες και την ημερομηνία έγκριση της έκθεσης. Οπότε πέραμε στην επόμενη φάση της συνεδρίασής μας, τις ψηφοφορίες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πόσες ψήφους έχει κάθε πολιτική ομάδα. Χαίρομαι που έχουμε αθρώα προσέλευση και τακτικών μελών και αναπληρωτών. Αλλά μην ξεχνάτε πόσοι, δικαιού, πόσοι ψήφους δικαιούται η κάθε ομάδα. Το ΕΛΚ 12, οι σοσιαλιστές 11, ή μάλλον λάθο, διορθώνει ο πρόεδρο. 13 ψήφου δικαιούται το ΕΛΚ και 12 οι σοσιαλιστέ. Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε αυτού του αριθμού. 13 ψήφοι για το ΕΛΚ και 12 για του σοσιαλιστέ. Γιατί βλέπω ότι έχετε περισσότερου ε, ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Δεν δικαιούνται όμω όλοι να ψηφίσουν. Yes, we we begin now with the πρώτη ψηφοφορία. για τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκεκριτής είναι ο κύριος Νταν Νίκα. Αρχίζουμε. Παρακαλώ. Είστε έτοιμοι. Ξεκινούμε. Τροπολογία 8. Ζητήθηκε από τον εισηγητή η υποβολή προφορικής τροπολογίας. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Συμφωνείτε με την προφορική τροπολογία του εισηγητού. Μήπως ο εισηγητής θέλει να πει κάτι. Την έχω υποβάλει και γραπτός, οπότε μπορείτε να τη διαβάσετε. Ωραία. Ψηφίζουμε τώρα τροπολογία 8 με την προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. <coughs> Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Α, συγγνώμη, διορθώνει η πρόεδρος. Τροπολογία 19. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Συγγνώμη. Είναι προφορική τροπολογία, οπότε πρέπει να ρωτήσω αν κανείς έχει αντιρρήσει. Ωραία. Τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 19 μαζί με την προφορική. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται και ευχαριστώ που με διορθώσατε. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 34 ψήφισαν υπέρ, δύο κατά και μία αποχή. Οπότε εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κύριε Νίτσα. Επόμενο. Κύριε Φανίστερο, θα θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να κάνω δύο-τρία σχόλια, αν μου επιτρέπετε, γιατί... Γιατί ήταν πολύ σύντομο το χρονοδιάγραμμα και δεν είχαμε πολύ χρόνο και πρέπει να δουλέψουμε στα αγγλικά και με υποστήριξαν πολύ οι από τις διαφορε ομάδες για να πετύχουμε τους συμβιβασμού που πετύχαμε. Βασικό στόχος των συναδέλφων είναι να υπάρχουν κοινή αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών μέσων αυτών. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι επιτροπή που το ψηφίζουν αυτό. Η ΕΚΟΝ και οι άλλες επιτροπές ακόμα εξετάζουν την έκθεση Μπούλμαν και Φερνάνδες. Η Επιτροπή Προπολογισμού και Ελέγχου Προπολογισμού. Θα δούμε τι θα γίνει και Αυτό ως γενική παρατήρηση. Φυσικά λοιπόν ε, πρέπει πολύ γρήγορα να εργαστούμε και μία από τις προτάσεις μου είναι να δούμε στη συζήτηση αυτή τι μπορούμε να εισαγάγουμε σε αυτό το επίπεδο. Έκανα λοιπόν μία πρόταση σε πρώτη φάση, στην πρώτη συνάντηση με την Κωνσταντ εκρελ καταλήξαμε σε μια σαφή, σε ένα σαφές ε, συμπέρασμα ότι δεν είναι σωστό να ανοίξουμε τους ε, εθνικούς φακέλους στη συνοχή, γιατί πρόκειται για ένα βασικό θέμα ότι η πολιτική συνοχή είναι στα χέρια των εθνικών κρατών και αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αλλάξει, ούτε καν να συζητηθεί στη συνέχεια πέτυχα ένα σεμιμαστικό κείμενο. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλες τις ε, δυνατότητες και αυτό προβλέπεται σε προφορική τροπολογία. Έδωσε το κείμενο για να το εξετάσουμε. Και το βασικό μήνυμα είναι ότι καλό είναι να υπάρχει πιο ενεργή προσέγγιση από πλευρά τη Επιτροπή μα και αν είναι δυνατόν. Uh, στο τέλος τη περίοδου 2018-2020 να δούμε τι θα κάνουμε με το εργαλείο αυτό. Εμείς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως Κοινοβούλιο δεν ήμασταν καθόλου ικανοποιημένοι με την αφαίρεση κοντελίων από το γράμματά μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που ήθελα είναι να εξετάσουμε από νομικής άποψης τις δυνατότητες στην επερχόμενη συζήτηση να δούμε τι θα γίνει με το αποθυματικό απόδοσης. Να σας πω ότι πολλά καλά πράγματα πετυχαίνουμε με την πολιτική συνοχή, με το ERDF και στις ε, αντιπροσωπείες μας ε, έχουμε σκεφτεί πολλά από τα τεχνολογικά αυτά, από τις τεχνολογικές αυτές εγκαταστάσεις και είναι πολύ ακριβά και μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνουμε ότι είναι μισοάδειες ε, γιατί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα εντάξουν αυτά στον τρόπο εργασία τους, στο σύστημά τους. Και το νέο χρηματοπιστωτικό εργαλείο δίνει ορίζοντα σε κάποιες περιπτώσεις 10-20 χρόνων. για να υπάρχει καλύτερος αντίκτυπος στην πραγματική ε, οικονομία. Άρα έχουμε αφενός ε, τα περιφερειακά κονδύλια και αφετέρου την κρίση και την ανάκαμψη μετά την κρίση. Γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση προτείνω να ψηφίσουμε και θα σας πω σε ποιο σημείο στον εκλογικό κατάλογο, στον κατάλογο ε, Τη ψηφοφορία θα φτάσουμε εκεί, να, να ψηφίσουμε και να μπουν αυτά τα στοιχεία στις συλλογικές σκέψεις, όχι όμω στο διδακτικό. Αποσύρω το κείμενο από το διδακτικό στην πρόταση. Να υπάρχει η βασική ιδέα και πρόεδρε να κλείσω λέγοντα το εξή. Τώρα θα πρέπει να γίνει αυτό, αναρωτιόμαστε. Όχι, όχι απαραίτητα ίσως, αλλά Το κάναμε και στο παρελθόν, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση. Η Επιτροπή μας ε, υπέβαλε κάποιες ιδέες και το Κοινοβούλιο το έβαλε και μέσα στις συνθήκες για τις συνέργειες. Το κείμενο αυτό λοιπόν το υιοθέτησε τελικά από το Κοινοβούλιο και στη συνέχεια το Συμβουλίο. Γιατί λοιπόν να καταθέσουμε μια ιδέα, θα το βάλω ως προφορική τροπολογία στον κατάλογο των ψηφοφοριών και σας δώσω την υποστήριξή σας. Once again. Thank you. Thank you for this extension. Η Πρόεδρος. Ε, δεν θα ήθελα να συνεχιστούν οι συζητήσεις. Α, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες λοιπόν στο σημείο αυτό. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με εισηγητή τον κύριο Φανίστεροι. Συμβαστική πρόταση υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, εγκρίνεται. Η 86. Τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 4 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 4 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά άποχες Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 105. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. 110. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Το πρώτο τμήμα μόνο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα περνάμε στην 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Η 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 102. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα της 102. Τρίτο τμήμα της 102. Υπέρ. Μάλιστα. Ακούω ότι υπήρξαν αλλαγές και οι αλλαγές ε, απεστάλησαν προς τις πολιτικές ομάδες χτες, ίσως και μετά χτες αργά το βράδυ. Πολύ αργά το βράδυ. Έχουμε λοιπόν την αλλαγή αυτή. Θέλετε χρόνο να διαβουλευτείτε πολιτικές ομάδες. η ε, κυρία Κρέλ. Τι ψηφίζουμε όμως τώρα, γιατί νόμιζα ότι έχουμε τον τελικό οριστικό κατάλαβο. Το τρίτο τμήμα, λέει ο Πρόεδρος, της τροπολογίας υπαριθμών 102. Στην παράγραφο 3. Α, πεστάλη χθες αργά το βράδυ. Να επανέλθουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Τρίτο τμήμα της 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ρεπετέ. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 154. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Πρώτο βήμα. Έχουμε ψηφοφορία σε δύο, τρία τμήματα. Δύο τμήματα βασική 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Δύο ψήφοι υπεράριθμες από τους σοσιαλιστές. Πέρας ψηφοφορίας και θα ξαναψηφίσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε αναπληρωματικά μέλη στην αίθουσα. Σας παρακαλώ μην ψηφίζετε. Να μετράτε πόσοι ψηφίζετε. Ας ελέγξουμε λοιπόν τώρα την 156 ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 37 ψήφοι, 19 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται η ψηφοφορία. Η τροπολογία. Και τώρα περνάμε στην 157. Υπέρ. Υπέρ της 157. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 157. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα ψηφοφορίας. Πέρας. Ίδιο το αποτέλεσμα. 20 υπέρ, 19 κατά. Άρα, η τροπολογία εγκρίνεται. Η 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα είναι σαφές ότι απορρίπτεται. Η 14. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Την τροπολογία 14. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Η τροπολογία περνάει. Έγκρινεται. 15, τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 166 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στην ανθρωπολογία 16. Υπέρ. Κάθα. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 17. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε, έναρξη της ψηφοφορίας, ψηφίσετε. Πέρασε. Είκοσι δύο ψήφοι 10 17 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Και συνεχίζουμε με την συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Η 20. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Η εννέα. Συμβαστική εννέα. Υπέρ. Κάτα. Άποχες. Έγκρινεται. Η συμβαστική δέκα. Υπέρ. Κάτα. Άποχες. Έγκρινεται. Η τριάντα. Τριάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ε, συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 31. Α. Καταπίπτει 31 επειδή δεν εγκρίθηκε η τροπολογία 86. 36 κατά πίπτη επειδή ούτε η 89 εγκρίθηκε και ε, πάμε στη συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Η 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 14. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 55. Η 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την τροπολογία 55. Ηλεκτρονικός έλεγχος έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισε τώρα. Ψήφισε τώρα. Πέρα της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 15 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 59. Ε, 59. Υπέρ. Κατά με αποχές απορρίπτεται. Σεμιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σεμιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17. 17. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 70. Υπέρ. Κατά αποχές. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, παρακαλώ, για την τροπολογία υπαριθμών 70. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Δεκαεννέα ψήφι υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. σε 73. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Κρέλ. Κάτι για το 75 θέλω. Είμαστε στο 73 ακόμη λέει ο πρόεδρος. Να κάνουμε το 73 και μετά πάμε στο 75. 73, there is an oral amendment. Στο 73 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση κατά της προφορικής. Όχι. Και τώρα ψηφίζουμε την 73 με την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίνεται. 74. We go. 74. Α, ναι, ναι, ναι. την ναι, ναι, ναι. Πάμε στο 75, συγγνώμη λίγο. Και εδώ έχει ζητηθεί ε, προφορική τροπολογία. Είναι κανεί κατά τη προφορική. Κρέλ. Οπότε, κατάλαβα τι είπε ο Σιθής στην αρχή, αλλά όμως Ήδη υπάρχει ένας εθνικός φάκελος στην ε, πολιτική συνοχή και λόγω της χρονικής εστέρησης θέλω να του ζητήσω να ε, αποδεχθεί προφορική τροπολογία επί της προφορικής τροπολογίας. Είναι πάρα πολύ απλό. Σας θα διαβάσω το κείμενο. Ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στην αρχή του προπολογισμού στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιτού πλαισίου του δημοσιονομικού κάποια ε, εγγύηση για προγράμματα πέραν του ορίζοντος 2020 και του Connecting Europe Facility. Νομίζω ότι έτσι τα καλύπτουμε όλα και είμαστε ίδιο μήκος κύματος, αλλά όμως δεν, έτσι φεύγει η δυσκολία ε, που έχουμε ίσως περιφερειακή για την περικοπή των κονδυλίων της ε, πολιτικής συνοχής. Ελπίζω η πρόταση αυτή να βρει υποστηρικτές. Okay, we have checked. Πρόεδρος. Έχουμε επομένω δύο προφορικέ τροπολογίε τώρα. Για να δούμε τώρα αν θα αποδεχθεί την πρόταση ο κ. Φανίστελβα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πέστε μας. Ναι, τώρα μου το κείμενο. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ανοιχτή προσέγγιση για καλυφθούν όλε οι πιθανότητε όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση σε σχέση με τι εγγύσει για το Connecting Euro Facility για το Horizon. Όμω κρίμα που σε αυτό το κείμενο δεν αναφέρεται το θέμα των επιδόσεων ρητός. ήθελα να πω στην κυρία Κρέλ ότι στην συζήτηση θα πρέπει να περιλάβουμε τις επιδόσεις, τις, τους περιορισμούς και λοιπά όπως εξήγησα. Και να δούμε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα να καλυφθεί και το θέμα αυτό των επιδόσεων. Εσείς με αυτή την ε, διατύπωση δεν, το, δεν τις αποκλείετε. Όχι, δεν τις ε, αποκλείω, λέει η κυρία Κρέλ, γιατί λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται κάτι να μας, ε, να μας παραδώσει, να μας διαβιβάσει σε σχέση με το ορίζον 2020 και για τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΙ, του ΕΤΣΙ τέλο πάντων και αυτά, αυτά ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, ο εισηγητής σας ε, δεν είναι για τόσο ενθουσιασμένος από όλα αυτά, αλλά διαπιστώνει ότι μπορεί να επαναφέρει τις ε, προτάσεις του τότε. Μια που έχουμε μια διαδικασία κατά κάποιο τρόπο εξαιρετικού χαρακτήρα. Και τέλος πάντων αποδέχομαι την ε, τροπολογία ως συμβασμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πρόεδρος, πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε πνεύμα συμβαστικό διότι θα υπάρξει ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Επιτροπή μας παρουσιάσει την ε, ε, αναθεώρηση αλλά και όσον αφορά το αποθεματικό επίδοση. Εντάξει, θα το περιλάβουμε, λέει ο κ. Άρα τώρα έχουμε να ψηφίσουμε αυτή την μία προφορική τροπολογία που έγινε αποδεκτή. Θέλετε το λόγο. Ναι, ναι, θα θέλαμε όμω να δούμε το κείμενο, να δούμε το έγγραφο γιατί το κόμμα μα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τι θα ψηφίσουμε εξαρτάται απολύτω από αυτή τη διατύπωση. Εγγράφο παρακαλώ. Θέλετε λίγο χρόνο για να το διαβάσετε. Okay, this is really a crucial moment in, in the vote. So. Πολύ σημαντικό σημείο τη ψηφορία. We can have one minute. Ένα λεφτά για να σας δώσουμε, λέει ο κ. Φανίστερ. Ναι, ναι, ναι, ένα λεπτό για να διαβάσετε το κείμενο. Okay. Thank you. One minute is gone. Πέρασε τον ένα λεπτό, λέει ο Πρόεδρο. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Do we have any other Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα? Όχι, απλώς είναι θέμα πειθαρχίας. Καθίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους και έχουμε μόνο αυτή την προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι κατά της προφορικής. Όχι. Σας ευχαριστώ. Επομένως, ψηφίζουμε τώρα. Το 75 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Και εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 76. Τι είναι υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Απαλήθευση για το 76 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Τώρα. Πέρα της 18-21. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Συμβεστική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το ναι, να ψηφίζουμε. Πέρας. You didn't vote? Oh. Δεν ψηφίσατε. Okay. I Can we Can we it is it will be e- Πρόεδρος. Καλύτερα να επανελθεί η ψηφορία. Άρα, καταπίπτει η προηγούμενη ψηφορία και θα επαναλάβουμε την ηλεκτρονική ψηφορία επί του 81. 81 ηλεκτρονικά. Τώρα. The vote is closed. Πέρασε ψηφορίες. Το εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τώρα. Πέρας. 32 δύο υπέρ. Έξι κατά. Ευχαριστούμε εισηγητά και ευχαριστώ όλους. Και ευχαριστούμε για τους συμβασμούς. So, the next vote... Η επόμενη ψηφοφορία. Είναι ε, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για στρατηγικές ε, επενδύσεις. Συγχαρητήρια ο κύριος Φαν Νιστελρόη. Δεν έχουμε κάποια άλλη παρατήρηση και αρχίζουμε την ψηφοφορία. Ξεκινούμε με την ε, τροπολογία υπαριθμών 1. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολόγη υπερθυμών 2. Έχει αποσυρθεί. Λόγω της πρώτης και πάμε τώρα στην υπερθυμών 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Καταπίπτει. πέντε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. απολύτως, έξι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Για την τροπολογία υπαριθμών 6 ψηφίσμα. Πέρας. Δεκανέα είκοσι. Απορρίπτεται. Επτά, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορείτε να πάμε στο εννέα, υπέρ. Κατά. Αποχέ Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Με την προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική. Όχι. Επομένως ψηφίζουμε για το 14 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφορία τώρα. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Τριάντα πέντε. Εγκρίνεται η έκθεση. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια κύριε εισηγητά. Η επόμενη έκθεση. Επόμενη ψηφοφορία. Έχουμε μία και μόνη ψηφοφορία. Αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 13-11 ε, του 2013 για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ε, περίοδο 14-20 μία και μόνη ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα Πέρας. Τριάντα εννέα. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πρόκειται το, τώρα έχουμε το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 2. Δεν έχουμε κάποια παρατήρηση και αρχίζουμε τώρα. Με το πολύ υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την τροπολογία παριθμών 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. 18-20. Η τροπολογία 3 απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμόν 1. Χωριστή ψηφοφορία. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Συμπαθάτε με λέει πρόεδρος γιατί Κάτι ξέρασα. Δεν είδα το σύνολο του κειμένου. Έχουμε και μια προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Επομένω. Το πρώτο τμήμα τη συμβασίας τροπολογία παραθυμών 1 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Τι συμβαστική. και το λόγο. Πώς αφού το πρώτο που λέει αυτές τις προσπάθειες και μετά πάμε στο δεύτερο τμήμα σε σχέση με αυτά που γράφει. Στο πρώτο τμήμα δεν υπάρχει αυτή η φράση. Στο δεύτερο, το δεύτερο, δεύτερο τμήμα είναι με αυτές τις λέξεις. Πρόεδρος. Είναι διαφορετικά κομμάτια. Ε, πρόκειται για την ίδια φράση, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικό τμήμα της. Ε, τροπολογίες. Οπότε τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής παριθμών 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. Και πάμε We go now to amendment 4. Uh, who is in favor? Πάμε στο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Του πρώτου υπαρθμών 5. Χωριστή ψηφορία εις δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κρέλ, ε, αυτό έχει καλυφθεί από τον συμβασμό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα του 5. Συμπαθάτε με, λέει η κυρία Κρέλ. Έχετε, έχετε δίκιο, λέει η πρόεδρος. Ε, δεν είναι σωστή η λίστα ψηφοφορία που έχω. Άρα, το 5, 6 και 7 αλλά και το 8 καταπίπτουν. Γιατί ενεκρίθη η συμβαστική παρθυμονένα. 1. Οπότε πάμε τώρα στην Τροπολογική παρθυμονένα. 9. Τι είπατε, έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί, ωραία. Και πού πάμε στη Συμβαστική Παριθμών 2. Έχει σφάλματα η κατάλληλη που έχω Και το πάμε τώρα. Στη συμβαστική υπαριθμών 2 είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και πάμε. Στην 12. Υπάρχει έτοιμα προφορική τροπολογία; Είναι κάποιο κατά? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία παραθμών 12 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Δεν κρίνεται. Τελική ψηφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Τριάντα ψήφια πέρα. Κανείς κατά. Ευχαριστώ. good job with... Έχουμε άλλες Όχι, α, θαυμάσια. Μπράβο μας. Κύριε Μποστινάρο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη συνεργασία που είχαμε και τη συνεισφορά σας. Και παρόλο που είχαμε συνοπτική διαδικασία και μεγάλη σπουδή, καταφέραμε εγκαίρως να εγκρίνουμε τις εκθέσεις. Και εγώ ευχαριστώ θερμά και τον εισηγητή και τους συνεισηγητές ε, γιατί ήταν πραγματικά δύσκολο του πιεστικού χρονοδιαγράμματος. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και για τη συμμετοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ανταλλαγή απόψεων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά προγράμματα και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Κατευθυντήριε γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Η συγγετής μας είναι ο κύριος Μπλάνκο Λόπες. Είναι παρόντες και συγητές και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τους ακούσουμε μετά τον εισηγητή όμως. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Λόπες. Παρακαλώ Όσοι αποχωρείτε από την αίθουσα, κάντε το αθόρυβο. Ο κύριος Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όντως, ε, αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί της εκθέσεως που θέμα έχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της μακροαιρεσιμότητας του άρθρου 23 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων. Θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι, μάλιστα ιδιαίτερα όσοι συμμετείχαν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, η οικονομική μακροαιρεσιμότητα ίσως είναι το πιο επίμαχο σημείο του κανονισμού περί κοινών διατάξεων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Η συγκεκριτής ήταν ο συντονιστής του ΕΛΚ, ο κ. Βανίστερ Ρόι, από κοινού με την συντονίστρια των σοσιαλιστών, την κυρία Κρέλ. Εξετάζοντας την έκθεση βλέπω ότι οι προτάσεις των συνεισηγητών του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών ήταν η ολοσχερής κατάργηση του άρθρου 23 του ΕΛΟΓΟ κανονισμού. Επιπλέον, διαβάζοντας τις τροπολογίες που, έχουν υποβληθεί εν ώψη της Ολομέλειας, βλέπω ότι η ολοσχερής κατάργηση του άρθρου 23 ε, ζητάται και με τις τροπολογίες της ΓΚΟΕ και των Πρασίνων. Οπότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ζήτηση που έγινε τότε για το άρθρο 23 έβρισκε απόλυτα σύμφωνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Βέβαια, οι ψηφοφορίες τότε δεν είχαν ε, ψηφιστεί και οι προηγούμενοι εισηγητές ε, της έκθεσης για τον κανονισμό γνωρίζουν καλύτερα από μένα τι έγινε με το κείμενο που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση από το Συμβούλιο και την Επιτροπή και στο οποίο εξακολουθούσε να περιλαμβάνεται το άρθρο 23. Βέβαια, ένα τμήμα της ιστορίας δεν φαίνεται στα, στα έγγραφα και μπορούμε να το φανταστούμε. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κατά της κατάργησης του άρθρου 23. Γι' αυτό και παρέμεινε το άρθρο στον κανονισμό. Ίσως όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τότε θα μπορούσαν να μας υπενθυμίσουν τι συνέβη. Εν πάση περιπτώσει, η μακροαιρεσιμότητα ήδη περιλαμβάνεται στον κανονισμό. Αποτελεί τμήμα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και δυστυχώ με την έκθεση τη πρωτοβουλίας στη δικιά μας δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Απλώς μπορούμε να επιδιώξουμε να εφαρμόζεται η μακροαιρεσιμότητα με τον πιο λογικό και ισορροπημένο τρόπο. Οι κατευθυντήριε γραμμέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι και το αντικείμενο τη έκθεσή μου, αφορούν το πρώτο τμήμα του άρθρου 23 δηλαδή μόνο τον αναπρογραμματισμό των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Και δεν αφορά το δεύτερο τμήμα του άρθρου 23, δηλαδή την διακοπή κονδυλίων. Είχα συνομιλίες και με μέλη της Επιτροπής και με σκιώδης ηγητές και εξοικειώθηκα με τις ανησυχίες τους. Επίσης συναντήθηκα με τις επιτροπές, με εκπροσώπους επιτροπών που θα γνωμοδοτήσουν. Και μάλιστα συνάντηθηκα και με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με εκπροσώπους ε, της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, μάλιστα, ο εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών θα έρθει το Μάιο στη συζήτηση της ε, έκθεσης. Πάντως, διαβάστε την έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες του αναπρογραμματισμού των ε, ταμείων και ποιο θα είναι το διοικητικό κόστος και η διοικητική επιβάρυνση αυτού του αναπρογραμματισμού. Γιατί μπορεί να επηρεάσουν ε, τις περιφέρειες, ε, τους δήμους και τις κοινότητες. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνηση, αλλά και διάφορες πτυχέ των αρχών της διαφάνειας και της διοργανικής συνεργασίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η οικονομική μακρο... μακροαιρεσιμότητα θα πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο την ε, εφαρμογή μιας βιωσιμότερης και αποτελεσματικότερης πολιτικής συνοχής. Δεν μπορεί η για να, χρησιμοποιηθεί για να πληγούν οι πιο υπερχρωμένες ε, περιοχές και περιφέρειες που εξαιτία της δινής οικονομικής κατάστασης ε, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις θα πρέπει περιφέρειες ε, ή τοπικές αρχές ε, να μην παραλύσουν εξαιτίας ενός αναπρογραμματισμού και λόγω της μη των μακροοικονομικών κριτηρίων που αντιστοιχούν σε κεντρικό επίπεδο διακυβέρνησης. Εξού και η ανάγκη ε, μέγιστου διοργανικού συντονισμού και διαθεσμικού συντονισμού σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης και αποφυγή της αποεθνικοποίησης, ε, ε, της επανεθνικοποίησης μάλλον, ώστε να μην διακυβευτεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που είναι ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Πάντως, ε, με προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο αναμειγνύεται η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι ο μοναδικός Θεματοφύλακα τη ε, σωστή εφαρμογή μακροαρισιμότητα είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεσή μου στο θέμα αυτό, τη σωστή συμμετοχή και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί, επαναλαμβάνω, έχει θεμελιώδη σημασία. Δεν θα αναπτύξω λεπτομέρειες, τώρα εκπονώ το σχέδιο της έκθεσης, γι' αυτό και περιμένω τις προτάσεις των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής. Θα στείλω το έγγραφο για μετάφραση μέσα σε δύο εβδομάδες, ώστε να μπορέσουμε στην επόμενη μας συνεδρίαση του Μαΐου να εξετάσουμε το έγγραφο και να, την ψηφίσουμε, να, να την έκθεση τον Ιούλιο μετά την κατάλληλη διορία για την κατάθεση τροπολογιών. Περιμένω λοιπόν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις εκείνων με τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μέχρι στιγμής. Με την ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να βρούμε τα κοινά μας στοιχεία, τον κοινό παρανομαστή, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνενετική έκθεση, η οποία δυνατό θα υπερψηφιστεί από την συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα θα έχουμε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για παρουσίαση ιδεών, προκειμένου να τεθούν οι προϋποθέσεις για την ανέβρεση μεγαλύτερης δυνατής συνένεσης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπλάνκο Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους και Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του εισηγητού μας, του κυρίου Λόπες. Όντως συναντηθήκαμε μαζί του, είμαστε σε επαφή συνεχώς και συμφωνώ με αυτά που είπε για το άρθρο 23 όλο το υπόβαθρο που μας περιέγραψε είναι σωστό, ισχύει. Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ανέβρεση συμβαστικής λύσης, ε, η δημιουργία συνένεσης. Και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε καλύτερα αυτό το άρθρο που ήδη υπάρχει στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Δυστυχώς ε, το περιθώριο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ περιορισμένο. Και από με την Επιτροπή Περιφερειών πιστεύουμε ότι το άρθρο 23 μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα και αρνητικά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους τοπικούς και περιφερειακούς φόρους. Γιατί η έκτη έκθεση περί συνοχής μιλά για υψηλό επίπεδο χρέωση, για υπερχρέωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά τη διακυβέρνηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή Περιφερειών αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν αλλάξει από τους αρχικούς προσανατολισμούς, αλλά δυστυχώς η σαφήνειά τους δεν έχει βελτιωθεί. Οπότε η Επιτροπή Περιφερειών ζητά περισσότερη προβλεψιμότητα και μεγαλύτερη σαφήνεια στη διατύπωση των κατευθυντηρίων γραμμών. Πάντως, επαναλαμβάνω, τα περιθώρια είναι στενά. Και όπως είπε ο εισηγητής μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαφυλάξει την ανάμειξή του και το ρόλο του Κάτι που περιμένουν από εμά και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και η Επιτροπή των Περιφερειών. Θα πρέπει να βρούμε σωστό τρόπο για να ερμηνεύσουμε το άρθρο 23. Συμφωνώ ότι το πρώτο σκέλος, το, το πρώτο τμήμα του άρθρου 23, ο αναπρογραμματισμός, περιλαμβάνει νέες διοικητικές επιβαρύνσεις και επιτείνει το διοικητικό φόρτο, κάτι που είναι αρνητικό. Επίσης, ε, δεν αναφέρεται με σαφήνεια κατά πόσο τα κριτήρια που αναφέρονται είναι ενδεικτικά ή όχι. Ή, θα πρέπει, ο κατάλογος των κριτηρίων είναι εξαντλητικός. Επίσης, μερικές διατάξεις ε, είναι ασυνάρτητες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα αιτήματα αναπρογραμματισμού μπορούν να υποβληθούν μόνο το 2015. Δεν έχει νόημα πια αυτή η διάταξη, γιατί είναι παροχημένη. Συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανοιχθεί στην όλη διαδικασία και να ασκήσει το καθήκον δημοκρατικού ελέγχου που έχει. Η παράγραφος 15 του άρθρου 23 θα πρέπει να διατυπωθεί με πιο διεξοδικό τρόπο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεόντως. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενισχυθεί η σχετική παράγραφος, ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να επιτελέσει απρόσκοπτα το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου του. Είναι σημαντικό το μέσο που προσφέρεται με τον κανονισμό αυτό, αλλά χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές για να το, εφαρμόσουμε, για το εφαρμόσουμε σωστά. Και παραλαμβάνω, οι γραμμές χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές. Έχω και μία ερώτηση. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ελλάδα ή τη Γαλλία. Πώς θα εφαρμόσει τη μακρορεσιμότητα στις δύο αυτές χώρες. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τι διαδικασία θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, δεν θα πρέπει η διαδικασία να επηρεάζεται από πολιτικές σκέψεις και να πολιτικοποιείται. Αυτά και ευχαριστώ τον εισηγητή μας για τη συνεργασία που είχαμε. Συνεχίζουμε με την σκιώδη συγγήτρια την κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ. Καλή είναι η οικονομική διακυβέρνηση και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση είναι σημαντική για τη σωστή εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής αλλά και για την ανάπτυξη σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σίγουρα θα πρέπει ε, τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση να τη χρησιμοποιήσουμε ως ε, τρόπο διεξόδου από την κρίση και αποτελεσματικότητα της οικονομικής ανάπτυξης προκειμένου να διορθώσουμε αρνητικές οικονομικές ε, προοπτικές όπως είναι η διαδικασία υπερβολικού χρέους ή υπερβολικό δημόσιο χρέος που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Το, ε, η έκθεση του 2013 φαίνεται ε, κατηκνύει μία διεύρυνση του χάσματος ε, και επιβάλλει ε, την, την ανάγκη τα προγράμματα να λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά διαρθρωτικά προγράμματα και τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα, καθώς και την εφαρμογή μέτρων με τα οποία εξασφαλίζεται η στήριξη ε, θεμελιωδών οικονομικών πολιτικών από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Εγώ είμαι υπέρ της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφεύγεται ο συχνός αναπρογραμματισμός, γιατί έτσι εμποδίζεται η προβλεψιμότητα και θίγεται η αξιοπιστία των εταιρικών σχέσεων. Οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα ανανεώνονται κάθε χρόνο. Οπότε είναι δύσκολο να γίνονται προβλέψεις μακροπρόθεσμα με κάτι τέτοιο, αν λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συστάσεις αναχώρα. Θα πρέπει με πολύ ε, προσοχή να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Εξουσία της για τον αναπρογραμματισμό και να δώσει έμφαση στην ε, ε, σταθερότητα και όχι στον πολύ συχνό αναπρογραμματισμό. Με το συχνό αναπρογραμματισμό θα πληγούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που ούτως ή άλλως δεν ευθύνονται για το υπέρμετρο δημόσιο χρέος αλλά από το σύστημα δεσμεύονται για μια ισορροπημένη ε, χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ρεν. Ο κύριος Βαν Μίλτεμπερκ θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί όντω ο δικαστή τον σκιώδησε γιατί μα για το θέμα αυτό. Τον κύριο Ρεν. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη ότι ήταν υπέρμαχος ε, μιας διαφανούς ε, διαχείρισης των, των προγραμμάτων για τη μακροοικονομική ρεσιμότητα. Θέλουμε να συμπληρωθεί, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό το πρώτο βήμα των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά Λαμβάνοντα υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενημέρωση ε, των βήματων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά τον ορισμό των λειτουργικών προγραμμάτων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές ή τις αναστολές πληρωμών. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει στην πράξη, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, όπως λένε και οι Άγγλοι, στην ε, πράξη φαίνεται ποια είναι τα προβλήματα και αν πετύχουμε κάτι. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην πράξη, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα εγκρίνουμε ως κοινοβούλιο ή τι ενδεχομένω πρέπει να χτενίσουμε παραπάνω. Πρόκειται για τι κατευθυντήριε γραμμέ και νομίζω ότι σε ένα διαρθρωμένο διάλογο θα μπορέσουμε να επισημάνουμε τα στοιχεία αυτά που μας απασχολούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ευχαριστώ. ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Άντερσεν, θέλετε το λόγο. Το Κοινοβούλιο ήταν κάθετο κατά αυτής της ε, ε μακροαιρεσιμότητας και εμείς το ΣΥΝΦΕΝ είμαστε και εμείς κατά αυτής της μακροαρισιμότητας γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα ψαλιδίσει ακόμη περισσότερο την οικονομική μας κυριαρχία. Γιατί αυτό γίνεται. Παίρνουν την κυριαρχία και την παραδίδουν στην Επιτροπή και έτσι επιβάλλεται περισσότερη ε, λιτότητα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους πόρους για τις στρατηγικές επενδύσεις χωρίς όμως να πάμε σε κάποιους περιορισμούς και λιτότητα. Θέλουν να αποκλειστεί η συνδιαχείριση. Ε, πώς θα υπάρξει ο υπολογισμός του ελλείμματος. Χρειάζεται να γίνουν κρατικές επενδύσεις όμως η Επιτροπή δεν αφήνει τα κράτη-μέλη να εμπλακούν στο πλάνο Juncker. Θέλουν απλώς να ελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν περισσότερες κρατικές επενδύσεις σε όλες τις περιοχές. Στη Βόρειο Ιρλανδία το συμφέρει είναι κατά αυτών των αποφάσεων Έχουμε συνεχείς περικοπές των κονδυλίων και οπότε είμαστε κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται και στο Λονδίνο και στο Δουβλίνο αλλά και στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να συρρυκνωθεί αυτή η επίδραση της μακρορεσιμότητας σε επίπεδο ένωσης. Αναστολή τι σημαίνει για τα μικρά κρατημέλη και για τις ε, περιφέρειες που στηρίζονται σε αυτά τα κονδύλια. Είπαμε για ένα προγραμματισμό της ε, Σύμφωνης Εταιρικής Σχέσης. Αλλά τι θα γίνει με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Με αυτές τις αποφάσεις η δύσκολη κατάσταση θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Δεν νομίζω ότι η Επιτροπή μας θέλει μια τέτοια εξέλιξη. Thank you very much. And... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Κύριε Ροπέ, θέλετε το λόγο. Όχι. Καλώ. Κυρία Μάλετιτς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα και πολύ περίπλοκο. Χρήζει λοιπόν της πλήρους προσοχής όλων μας. Φυσικά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την λύση μια μόνο και μοναδική προσέγγιση, γιατί υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορούμε την ίδια λύση να την εφαρμόσουμε σε όλου. Μερικέ χώρε έχουν ε, εθνικά προγράμματα και αλλε περιφερειακά. Γιατί ε, μερικές χώρες έχουν υποβάλει μόνο ένα, δύο, τρία τέτοια προγράμματα, άλλε χώρε ε, εκατοντάδε. Είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια προσέγγιση για όλους. Ας μην ξεχνούμε επίσης ότι δεν εννοείται περιφερειακή ανάπτυξη αν ολόκληρη η χώρα αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικά προβλήματα. Μην περιμένετε περιφερειακή ανάπτυξη όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και στόχος της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση και τέτοιων προβλημάτων Οπότε στόχος μας θα, πρέπει να, θα είναι να δημιουργήσουμε πρόσφορο επιχειρηματικό περιβάλλον, ελαστική αγορά εργασίας, ε, ε, υγιή, δημόσια οικονομικά και φυσικά μία δημοσιονομική εξυγίαση φιλική προς την ανάπτυξη. Γιατί σε πολλές χώρες μέλη εξαιτία όλων αυτών ε, των μέτρων, ε, των δρακόντιων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίασης διακυβεύεται η ίδια εφαρμογή των προγραμμάτων της συνοχής. Οπότε θα πρέπει να βρούμε σωστές λύσεις και να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχής για να ε, διορθώσουμε προβλήματα οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, θα πρέπει να έχει κατά νου ότι δεν αρκεί μία ίδια λύση για όλους εξαιτίας των διαφορών που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη. Οπότε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε επιτυχώς τις κατευθυντήρες γραμμές, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την απλότητά τους, ε, την λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων μεταξύ των χωρών και επίσης ε, να μας επιτρέπει μια έγκαιρη αντίδραση, μια άμεση, ταχεία αντίδραση. Να μην διακόπτουμε ή να μην αναβάλουμε εφαρμογή τέτοιων ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν εφαρμοστεί κάποια μέτρα που προβλέπονται από τις ειδικέ συστάσεις ανά χώρα. Επίσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια προγράμματα τεχνικής αρρωγής, κάποια επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής αρρωγής και να μην αλλάξουμε όλο τον τρόπο λειτουργίας των θεματικών προτεραιοτήτων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και σε αυτή τη φάση ε, οι κατευθυντήριες γραμμές με τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί δεν μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει στο μέλλον να καταστούν πιο λειτουργικές και πιο εύχριστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον συνάδελφο για την έκθεσή του για ε, αυτή τη θεματική που είναι τόσο, τόσο, τόσο επίμαχη όπως ε, και η μακροεσιμότητα και είπαμε ότι στο κοινοβούλιο είχαμε πάρα πολύ δώσει μία μάχη για να μην υπάρχει μία τέτοια διάταξη. Και αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το διαβόητο άρθρο 23 ανησυχεί τις περισσότερες πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διασκέδασε αυτές τις ανησυχίες μας για την αναστολή των εκταμιεύσεων με κάποια λογική. Και πέρσι ο κύριος Χάνο πρώην Επίτροπος είχε πει ότι η εφαρμογή της μακροαιρεσιμότητας προβλέπεται σε περίπτωση κατά την οποία τα κράτη-μέλη επιμένουν να μην τηρούν τις οικονομικές συστάσεις. Οπότε τελικά ε, ε, αυτό είναι μια θεωρητική ρύθμιση. Έτσι τώρα θα τιμωρηθούν κάποιες περιφόρειες, περιφέρειες εάν δεν ενεργούν όπως πρέπει. Πρόκειται για ένα εργαλείο της πολιτικής συνοχής και της ε, επικουρικότητας. Αλλά έτσι θα πληγούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν έχουν τα μέσα της σχετικής κυβέρνησης αλλά επίσης συνταγματικά ε, είναι δεσμευμένα όσον αφορά τον προπολογισμό τους. Και οπότε θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με την Επιτροπή των Περιφερειακών για να δούμε τι θα γίνει με την γνωμοδότηση αυτή του Φεβρουαρίου του 2015. Οπότε στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου όσον αφορά την ευελιξία του προπολογισμού είχαμε πει ότι αυτό θα βοηθήσει σε κάποιες ε, επενδύσεις αλλά θα πρέπει να γίνει επαναπρογραμματισμός των διαθροτικών ταμείων για να ληφθούν μέτρα για όσους δεν τηρούν ε, ε, αυτά τα οποία πρέπει. Οπότε πράγματι τι είναι το άρθρο 23 και θα θέλαμε να είμαστε πιο ε, τολμηροί στην αντιμετώπιση μας στην Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο το λόγο για την συζήτηση αυτή. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο ή ΕΚΦΙΝ. Αποφασίστε μεταξύ σα. Έχετε το λόγο. σα ευχαριστώ πολύ από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε να ευχαριστήσουμε επίση και τους και και τον εισηγητή για τις διάφορες ε, παρεμβάσει που ακούσαμε σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω εξηγώντα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμέ. Η έγκριση των κατευθυντηρίων αυτών προέκυψε μετά από δήλωση στην ε, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διελευκάνει κάποια ζητήματα αναφορικά με την παράγραφο 1 έως 6 του άρθρου 33. Αυτό λοιπόν ήθελα να το διευκρινίσω, το άρθρο 23, συγγνώμη, ότι πρόκειται για διευκρίνηση των άρθρων των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 23. Η δήλωση λοιπόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει περαιτέρω την ιδέα της αναθεώρησης και το είδος των τροποποιήσεων και το τι θα μπορούσε να αποτελέσει δέουσα δράση όπως ορίζεται στην παραγραφό 6 να αναφέρει το είδος των συνθήκων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή των πληρωμών και τα κριτήρια τα οποία θα θεωρούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ισχύουν για να καθορίσει την αναστολή της ε, πληρωμής αλλά και το μέγεθο τη αναστολή, τη διάρκεια τη αναστολή. Αυτά λοιπόν τον Ιούλιο του περασμένου έτου αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν. Νομίζω ότι οι κατευθυντήριε γραμμέ λοιπόν απευθύνονται σε διάφορα ζητήματα τα οποία ήδη είχαν, έχουν οριστεί στι παρεμβάσει σα, Να διευκρινίσω το εξή ότι η συμφωνία και τα, προ... οι συμφωνίε και τα προγράμματα όταν εγκρίνονται θα πρέπει να αποκρίνονται στις συστάσεις του Συμβουλίου και στις συστάσεις αναχώρα. Θα πρέπει δηλαδή να συνάδουν με τις τελευταίες συστάσεις της γενικής οικονομικής πολιτικής. Αυτό, θα έχουμε υπόψη ε, ως πρώτο στοιχείο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που σίγουρα καθησυχάζει. Ελπίζουμε ότι τα προγράμματα δεν θα πρέπει σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον χρονικό ορίζοντα να τροποποιηθούν γιατί συνάδουν με τις βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής. Και ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό μόνο μεταξύ της περίοδου 2015 και 2019. Όχι λοιπόν τέτοια... Όχι το 2014. Επίσης, ε, τονίσατε στις κατευθυντήριες γραμμές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά τη σταθερότητα και όχι τόσο πολύ την ε, προγραμματική αναδιάθρωση, επειδή είναι δομικής και τεθοδικής σημασίας το στοιχείο αυτό και η πολιτική αυτή. Και σε περίπτωση αναπρογραμματισμού, αλλαγή των προγραμμάτων, αυτό θα λάβει χώρα μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος, δηλαδή ότι ή τα ωφέλη της αλλαγής των προγραμμάτων είναι πιο πολύ, πιο πολλά από τα μειονεκτήματα ενδεχόμενης αλλαγής των προγραμμάτων. Και σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των προγραμμάτων που θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αναφέρθηκε ότι πολλά, πολλές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη με τρία-τέσσερα προγράμματα μόνο σε όλη τη χώρα, ενώ άλλα κράτη-μέλη έχουν πολλά προγράμματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι η άσκηση αυτή θα πρέπει να παραμείνει όσο πιο απλή γίνεται. Και ο λόγος της διαφοροποίηση των κρατών μελών αποτελεί και την εξήγηση για το ότι οι κατευθυντήριε γραμμές δεν μπορούν να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί κάπου ασκήθηκε η κριτική ότι είναι πολύ γενικόλογε οι κατευθυντήριε γραμμέ και ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε επακριβώ πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει αυτή την αλλαγή των προγραμμάτων. Αλλά να θυμόμαστε, είναι πολύ σημαντικό ότι καταρχά ε, ο νομοθέτη αποφάσισε να δώσει κάποια διακριτική ευχαίρεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά δεύτερον δεδομένη τη τεράστια διαφορά, των τεράστιων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι κατευθυντήριε γραμμέ δεν μπορεί να απευθύνεται και να επιλύουν όλα τα ζητήματα και να είναι πιο συγκεκριμένε. Σε ό,τι αφορά την ιδέα τη αναθεώρηση και του τύπου των αλλαγών, αν υπάρχει σύσταση ανά χώρα ή σύσταση από το Συμβούλιο που έχει να κάνει που μάλλον ε, πρέπει να οδηγήσει σε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θα το πράξει αυτό μέσα σε 4-5 μήνες και θα αποστείλει την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη σωστή τεκμηρίωση στην πρόταση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα αναφέρει το ελάχιστο τις ελάχιστες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη, τον αντίκτυπο στην ε, χρηματοοικονομική διάσταση και τα προγράμματα και την προσδοκία ότι τα προγράμματα θα εφαρμοστούν. Θα ορίσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τομεί που θέλει να υπάρξει ενίσχυση. Αλλά θα επαφείτε, στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποια προγράμματα πρέπει να περιοριστούν για να αντισταθμίσουν το σύνολο. Γιατί αυτό συνάντηκε και με την αρχή της επικουρικότητας, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, μπορεί να τα ελέγχει όλα στην, ε, στο έτοιμά τη. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία δεν θα πρέπει να υποστούν μείωση. Επίσης, οι κατευθυντήρες γραμμές ε, ορίζουν το τι είναι αποτελεσματική δράση, παρατίθενται διάφορα στοιχεία. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβουν τα κρατημέλη στις προτάσεις τους, βάσει και των αντιδράσεων των κρατών μελών, θα εκτιμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα διάφορα στοιχεία τα οποία έδειξε και κατά πόσον υπήρξε απαρκής αντίδραση. Οι κατευθυντήριες γραμμέ επίση αναφέρονται στο θέμα των συνθήκων που ενδεχομένω να οδηγήσουν σε αναστολή πληρωμών. Προφανώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αντίδραση και απάντηση από πλευρά του κράτου μέλους. Ε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αναστολή των πληρωμών. σε περίπτωση που το κράτος μέλος επίσης ε, δεν αντιδράσει σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, τα προβληματικά. Ενδεχομένως να μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι να προχωρήσει σε αναστολή πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διακριτική ευχαίρεια να αποφασίσει κατά πόσον θα προχωρήσει σε αναστολή ή όχι. Τέλος δε, οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν και τα κριτήρια των προγραμμάτων που είναι υποψήφια προς αναστολή. Αυτό που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι θα ληφθούν υπόψη τρία κριτήρια. Η αναστολή θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και αναλογική για να δώσουν σωστά κίνητρα προς τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στα αιτήματα το, της Επιτροπής. Επίσης, δεύτερο κριτήριο, η ισότητα, η ίση μεταξύ των κρατών μελών και το μερίδιο του ΑΕΠ θα ληφθεί υπόψη και ότι ο δίκτυπος της αναστολής στο κράτος μέλος θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Και εδώ οι κατευθυντηρίες γραμμές ε, αναφέρουν ότι θα ληφθούν υπόψη και διάφοροι φορείς που ενδεχομένως να αλλάζουν τις ισορροπίες, για παράδειγμα, το κατά πόσο υπάρχει ανεργία, στο κάθε κράτος μέλος, ε, ε, οικονομική ύφεση και το καθεξή. Τέλο, να αναφέρω ότι ο λόγο για τον οποίο δεν αναφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι κατευθυντήριε γραμμέ είναι ότι αυτό αποτελούσε ένα από τα στοιχεία τη αρχική δήλωση ε, ήταν ξεκάθαρη η αρχική δήλωση σε σχέση με το τι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα σε ό,τι αφορά τις κατευθυντικές γραμμές, αλλά δεν υπάρχει, καμία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη και θα εφαρμόσει τα όσα προβλέπει παραγράφος 15. Θα συμμετέχει άμεσα το Κοινοβούλιο, άμεσα θα ενημερώνεται αν υπάρξει λόγος που ενδεχομένω να οδηγήσει σε αναστολή και σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεδεθειμένη να προχωρήσει στα πλαίσια διαρθρωμένου διαλόγου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Τέλος, να αναφερθώ σε κάποια από τα συγκεκριμένα σχόλια που έγιναν από πλευρά των βουλευτών. Για το διοικητικό άχθος, για παράδειγμα, ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προγράμματος, ακόμα και σε ελάχιστο βαθμό, θα σημαίνει επιπλέον γραφειοκρατικό άκτο και για την Επιτροπή και για το κάθε μέλο. Αλλά γι' αυτό λοιπόν αναφέρουμε ότι η αλλαγή προγραμμάτων θα γίνει μόνο όταν ο αντίκτυπο. Μόνο όταν τα ωφέλη είναι πιο μεγάλα από τα μειονεκτήματα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Νομίζω τα υπόλοιπα στοιχεία αναφέρθηκαν. Σε ό,τι αφορά την αναστολή. Και τον αντίκτυπο στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση. Να σα αναφέρω το εξή Η αναστολή δεν θα οφείλεται στο μέγεθος των οικονομικών προβλημάτων. Θα οφείλεται στην μη αποτελεσματική δράση από πλευρά των κρατών μελών. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτοί που διακινδυνεύουν αναστολή δεν είναι τα κράτη-μέλη που έχουν οικονομικά προβλήματα. Γιατί το βασικό στοιχείο είναι η μη αντίδραση από πλευρά του κράτου μελους όχι το μέγεθος του προβλήματος. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιδράει και θα απαντάει γρήγορα. Αυτό τέθηκε και στα ερωτήματά σα, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει άλλη επικάλυψη με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ελπίζουμε λοιπόν οποιοδήποτε έτοιμα αναπρογραμματισμού να έχει ολοκληρωθεί πριν ε, τι συστάσει αναχώρα του επόμενου έτου από πλευρά του Συμβουλίου. Αυτά προ το παρόν. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σα ευχαριστούμε. Πολύ διεξοδική η παρουσίαση που μας κάνατε και η εξηγήση που μας δώσατε. Από την ΕΚΒΗ, ΕΚΦΙΝ τώρα εκπρόσωπος. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ε, προτάσεις τους και τις παρεμβάσεις τους. Όπως είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, οι κατευθυντήριες ε, γραμμές αφορούν το πρώτο τμήμα ε, του μηχανισμού του άρθρου 23, δηλαδή τον αναπρογραμματισμό. Που θα επισέλθουμε σήμερα σε λεπτομέρειες για το δεύτερο τμήμα του μηχανισμού. Να σας θυμίσω κάποια γενικά σημεία της μακροαιρεσιμότητας. Καταρχήν, δεν είναι το άρθρο 23 που θίγει τις περιοχές, αλλά οι ε, κακές μακροοικονομικές πολιτικές. Αυτές είναι που θίγουν τις ε, πολιτικές, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε υγιή περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς ε, χρηστή μακροοικονομική διαχείριση. Από αυτήν την άποψη το άρθρο 23 είναι πολύ προσεκτικό και έχει λάβει υπόψη τις διάφορες ανησυχίες και τον προβληματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εκφράστηκε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Και στα δύο σκέλη του μηχανισμού προβλέπονται πολλές ασφαλιστικές κλίδες στην μακροαιρεσιμότητα. Τέλος, ό,τι αφορά την ε, μεταχείριση της σύγχρηματοδότησης στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, γιατί τέθηκε σχετική ερώτηση. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει πλήρως την ευελιξία που επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη για να επιτρέψει δημόσιες επενδύσεις με τρόπο βέβαια δημοσιονομικά υπεύθυνο και γι' αυτό στις 30 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της ε, με την προσέγγιση της. Ε, στόχος μας είναι να τονώσουμε την ανάπτυξη με δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο, επαναλαμβάνω. Οπότε η ανακοίνωση τώρα εξετάζεται στις αρμόδιες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και θα εφαρμοστεί σχετικά σύντομα. Σας παραπέμπω στην ανακοίνωση που βρήθη πληροφοριών. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την δική μας Επιτροπή, γιατί ουσιαστικά συνεχίζει το έργο της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Επίσης, θέλουμε να διατρανώσουμε το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής. Και θα εξασφαλίσουμε σωστό έλεγχο του συστήματος ώστε να γίνει ισότιμη μεταχείριση των περιφερειών και των κρατών για να υλοποιηθούν οι στόχοι τους στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Αυτή την επιτήρηση θα την εξασφαλίσουμε με αυστηρό τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τις σκέψεις τους και μιλάμε για το 23, αλλά το άρθρο αυτό τι λέει. Λέει για το πώς θα μπορούσε να γίνει κάποια ισόρροπη και δίκαιη, ισορροπημένη και δίκαιη εφαρμογή ε, των ε, προβλεπομένων Επομένως το θέμα είναι τώρα να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της ε, Επιτροπής της Περιφερειακής και να δούμε τι γίνεται ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτήν την μακρορεσιμότητα εδώ εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ όλους επομένως για ότι είπατε, θα ήθελα τώρα να επανέλθουμε για να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο το είπαμε στην αρχή. Γιατί με, ανησύχησαν αυτά που άκουσα τώρα στο τέλος. Και τι εννοώ. Βεβαίως και είναι δυνατόν να εξαρτηθούν οι επενδύσεις και οι πόροι των περιφερειών και των τοπικών αρχών από την ε, μακρορεσιμότητα και αυτό να εφαρμοστεί όταν υπάρχει κάποια κακή διαχείριση από ένα κράτος ή τέλος πάντων κάποια, κάποιο, ε, κάποιο φορέα. Οπότε γι' αυτό το λόγο μπορούμε να έχουμε αναπρογραμματισμό όταν δεν ε, τηρηθούν κάποιες υποχρεώσεις που έχουν αναλυθεί. Και επομένως δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης. Είναι δυνατόν να έχουμε ε, κάποια μη τήρηση υποχρεώσεων ε, και από την κεντρική ε, εξουσία. Επομένω, αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε είναι το πώς δεν θα έχουμε κάποιου είδους κυρώσεις που να μην είναι δίκαιες και τέλος όπως είπε κάποιος μίλησε να επιδεινώσουν κάποιες καταστάσεις που ήδη είναι άσχημες. Οπότε γι' αυτό έχουμε αυτή την έκθεση. Ε, να ότι είναι εξισορροπημένη και δεν αμφισβητούμε για αυτό το άρθρο, γιατί αυτό το άρθρο είχε εγκριθεί. Δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε τη ζήτηση. Θέλουμε να αναζητηθούν κάποιοι ε, μηχανισμοί, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να εγγυηθεί την εφαρμογή της αρχής της αιρεσιμότητας και αυτή η εφαρμογή να γίνεται με τρόπο δίκαιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε ε, τα όσα είπαν οι σκιώδες συζητητές και ε, έτσι σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε για τόσο σημαντικό και γι' αυτό και εγώ θέλω να υπάρχει αυτό το θετικό πνεύμα ε, και έτσι να συνεχιστεί αυτή η συνένεση μέχρι το τέλος διαδρομής της έκθεσης και τις επόμενες ε, ημέρες ε, πριν έχουμε την επίσημη ε, συζήτηση με τους ε, συζητητές θα τους πω τι έχει γίνει ώστε να μας πούν τις σκέψεις τους τόσο σημαντικές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Και τώρα, ολοκληρώσαμε τα θέματά μας για την πρωινή συνεδρίαση. Οπότε, σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε με τη συνάντηση των συντονιστών. Ας μείνουν επομένως στην αίθουσα οι συντονιστές και θα συνεδριάσουμε και κλεισμένο των θυρών. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι να έρθουν στις 3 η ώρα θα τα πούμε τότε.